Είναι ένα τεράστιο επίτευγμα και ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ και γι' αυτό. Με το Horizon Europe λοιπόν έχουμε στείλει ένα ηχηρό ε, μήνυμα στους διαπραγματευτές ε, του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου για την επιστήμη, την καινοτομία και τώρα είναι κοινό μας καθήκον να υπερασπιστούμε ε, το προπολογισμό για όλα αυτά. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και επιλογίζω σε εσά, σε όλου σα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι ορίζοντα Ευρώπη όχι μόνο θα γίνει το μεγαλύτερο ε, πρόγραμμα καινοτομία και επιστήμη που έγινε ποτέ, αλλά και ότι θα φέρει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα για του πολίτε μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον Επίτροπο και τώρα σας ακούσουμε τις ε, απόψει. Ε, Σάντσες Από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Ε, εμείς απέχουμε ε, έρευνα, ανάπτυξη θέλουμε, καινοτομία, αλλά δεν έχει αλλάξει ε, η, τακτική. Για ποιο λόγο το κάνουμε και για ποιον σε σχέση με τον παλιό ορίζον 2020. Επίσης, είναι σκανδαλώδης ε, εμπλοκή με την αρχή ε, της προφύλαξης. Εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε απερίφραστα με την οικολογική κρίση, την ε, ισότητα των φύλων, την απασχόληση, την πρόσβαση στην υγεία, την καταπολέμηση των αδικιών. Αυτό που θέλουν είναι να αποδίδουν οι επενδύσεις, οι δημόσιες επενδύσεις, οι ιδιωτικά ε, έργα. Για άλλη μια φορά η κερδοφορία είναι προτεραιότητα ε, και όχι οι άνθρωποι. Και επειδή είναι η τελευταία μου παρέμβαση θέλω να ευχαριστήσω τους ψηφοφόρους και τις ψηφοφόρους που το 2014 μου ε, έδωσαν την εμπιστοσύνη τους, την Αμέλεια, τη Βιβιάνα, τον Χάρλος, τον Ζαγκόπ, ε, την ε, Δαβίδ και άλλους ε, από τους Ποδέμους στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, γιατί αν δεν σας είχα εσάς δεν θα είχα φτάσει ως εδώ που είμαι. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε. Τόρβαλτς από την Επιτροπή Προπολογισμού. Παρακαλώ ένα λεπτό. Kiitos arvoisa Μερικές φορές οι εργασίες στην Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι λίγο βαρετές, περίπλοκες. Οι δομές ε, δεν είναι και τόσο διαφανείς μερικές φορές και όταν μιλάμε για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε όρους που χρησιμοποίησε ο Επίτροπος και οι πολίτες συχνά οδηγούνται να σκεφτούν ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό δεν είναι παρά μια μαύρη τρύπα και εκεί μέσα στην οποία χάνονται όλα τα κονδύλια. Γι' αυτό το λόγο ε, είδαμε μεγάλο ενθουσιασμό το ότι πετύχαμε όλα αυτά τα ποσά για, να, για τον ορίζοντα Ευρώπη και καταφέραμε να επιτύχουμε μια συνένεση. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε πολλά για να πείσουμε, διότι τα κονδύλια ήταν αναγκαία. Ίσως ε, σε μερικές δεκαετίες να μαζέψω τα εγγόνια μου και τα δυσέγγονά μου και να τους πω τι έκανε ο παππούς, ο προπάπους τους όσον αφορά αυτά τα δισεκατομμύρια τα οποία θα χρηματοδοτήσουν αυτές τις εργασίες έρευνα που είναι τόσο απαραίτητε για την Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Η κυρία Αντιλαμπαγιώβα από την Επιτροπή ε, Συνταγματικών Υποθέσεων. Ελέγχου του προπολογισμού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα ε, η παγκοσμιοποίηση ε, προχωράει και θα πρέπει εμείς να επενδύσουμε στην καινοτομία και στην έρευνα. Ε, δεν έχουμε πολύ ε, μεγάλη εστίαση εμείς σε αυτό. Ε, παρόλο που ο ορίζον 2020 έφερε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στην ανταγωνιστικότητα, στην καινοτομία, αλλά θα πρέπει να ενισχύσουμε τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων. Να συνεχίσουμε να πλουστεύουμε τους κανόνες και τις διαδικασίες. Επίσης, θα πρέπει να τα μεταφέρουμε όλα αυτά καλύτερα στους πολίτες. Ο Horizon 2020 έχει ενισχύσει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Ο Horizon Ευρώπη τώρα θα πρέπει να διαδεχθεί αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Ευχαριστούμε κύριε για Ένα λεπτό. Grazie molto, stimați colegi, programul Orizont Europa va fi cel mai ambițios program από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. θα είναι ε, το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα για την έρευνα και την γενοτομία Ορίζων Ευρώπη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές και τη Ρουμανική Προεδρία για την εξαιρετική ε, δουλειά. Εγώ είμαι ο συντάξης ρομοδότης της Επιτροπής ΕΝΒΗ Περιβάλλοντος. Η πρότασή μας για την καταπολέμηση του καρκίνου είναι η προτεραιότητα. Εγκρίθηκε και από το Συμβούλιο και χαίρομαι γι' αυτό. Επίσης, 35% του συνόλου του προπολογισμού, 120 δις, θα στραφεί προς την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Και αυτή ήταν δική μας σύσταση τη Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θέλω να ευχαριστήσω ε, του συναδέλφου που ε, αύξησαν τον προπολογισμό της υγείας από 7,7 σε 9,12 δισεκατομμύρια. Ε, ε, ιδιαίτερα για τις καινοτόμες λύσεις, για την ογκολογία, για την καταπολέμηση του καρκίνου. Αυτά θα είναι ζωτικά για τις επόμενες γενιές, γιατί έχουμε κάθε χρόνο 35.000 νέα κρούσματα καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την Επιτροπή Μεταφορών. Βίρκουνεν, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους της Επιτροπής Μεταφορών ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους ε, τους διαπραγματευτές ε, για την άριστη κατά την άποψή μας έκθεση για τις μεταφορές υπάρχουν τρεις σημαντικές πτυχές πρώτα απ' όλα πρέπει να αυξήσουμε το κονδύλιο έρευνας και ανάπτυξης ε, για όλα τα κράτη-μέλη και στον ορίζοντα 2020 για να φτάσουμε στα 120 εκατομμύρια ευρώ για τις μεταφορές αυτό είναι σημαντικό έτσι θα γίνει η βιομηχανία μας ανταγωνιστική στο μέλλον και θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις τεράστιες παγκοσμίες προκλήσεις. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Μεταφορών στηρίζει τους κλιματικούς στόχους στο πρόγραμμα έρευνας όσον αφορά την κυκλοφορία, τις μεταφορές, την ε, εγκατάλειψη των ανθρακούχων εκπομπών. Είναι σαφές ότι Χρειάζεται έρευνα στο, στο μισθό μεταφορών και μετά όσον αφορά τις μεταφορές δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο κλάστερ. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε το κλάδο εγκάρσια ούτω ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ενέργεια, το κλίμα, οι μεταφορές, ε, η ενέργεια ε, και η βιομηχανία από κοινού. Είναι σημαντικό να κοινοτομήσουμε θεμελιδώ σε όλου αυτού του τομεί. Ε, ευχαριστώ, κύριο Βανίστα Λερόι, για την Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εισηγητέ, καμπή πραγματική. Μετά από 15 χρόνια εργασίας στις Επιτροπές Ήτρε και Ρέγγι, ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα περιφερειακά ταμεία με τρόπο ε, πιο ευέλικτο, χωρίς κρατικές ενισχύσεις. Ανά κράτος μέλος. Και βλέπω τώρα ε, τον ορίζοντα 2020 ως το ε, ε, παγκόσμιο Airbus ε, και τουλάχιστον 5% είναι οι συνέργειες, αλλά θα μπορούσαν και πολύ περισσότερο. Και μετά, η προβολή, το Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε με την έρευνά του ότι εμείς δεν φτάνουμε στους πολίτες. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το πάρει αλλιώ για να φτάνει στους πολίτες, να αλλάξει τρόπο επικοινωνία για να προβάλλουμε και αυτά που κάνουμε. Let the stars shine. Να προβάλλουμε αυτά που κάνουμε και διεθνώς. Και τέλος. Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι έχουμε ε, ε, αποτελέσματα και το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο, το Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Συμβούλιο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο καλή συνεργασία. Η κυρία είναι από την Επιτροπή Γεωργίας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Το Horizon 2020 ε, θα είναι πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα ε, σε ολόκληρη, για ολόκληρη την ανταγωνιστικότητα της Υπήρου. Πρόγραμμα μέσω του οποίου η καινοτομία στην Ευρώπη και οι επιστήμες θα αναπτυχθούν σε παγκόσμιο επίπεδο ανταγωνιστικά με τη ΣΥΠΑ και την Κίνα για παράδειγμα ως ε, ε, η συγγήτρια της Επιτροπής Γεωργικών Υποθέσεων υπογραμμίζω πόσο σημαντική είναι η αγροδιατροφική αλυσίδα, τα δάση, τα εσωτερικά ύδατα τα υψηλά κονδύλια για να εγκαταλείψουμε τις ε, ενέργειες που βασίζονται σε ορεικτούς πόρους πρέπει να είναι πρωτοπόρος Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διατροφικής ασφάλειας και σε θέματα ε, χρήσης των πρώτων υλών. Όταν θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει και οι τριμερείς διάλογοι το φθινόπωρο ε, για το CFP θα πρέπει να φροντίσουμε όσα προτείνει η Κομισιόν αυτό το, η δέσμευση του 10% να ε, διατηρηθούν. Ροντρίγκε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ε, το πρόβλημα Horizon Ευρώπη είναι ένα πρόγραμμα για την απασχόληση, την ανάπτυξη, για μεγαλύτερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα για τις συνεργασίες με πανεπιστήμια, ευρωπαϊκά και μη. Οι νέοι ερευνητές θα πρέπει να ε, συμμετέχουν και να συνδιαμορφώνουν τον ευρωπαϊκό επιστημονικό και ερευνητικό χώρο για να αποφύγουμε και τη διαρροή εγκεφάλων. Επίσης θα πρέπει να έχουμε περισσότερη ε, σύγκληση ε, και ιδιαίτερα οι άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες που είναι και σε μειονεκτική θέση και σε μικρότερη ανάπτυξη θα επωφεληθούν ε, και θα υπάρξει καλύτερη διασπορά των αποτελεσμάτων της έρευνας και της επιστήμης. Επίσης, στην τεχνολογία και στη θεμελιώδη έρευνα πρέπει να κάνουμε περισσότερα και στις κοινωνικές επιστήμες, ε, λαμβάνοντας υπόψη πάντα και τον πολιτισμό, διότι κατά τα άλλα η ανθρωπότητα θα είναι κάτι το οποίο θα βλέπουμε υπερβολικά μονοδιάστατα. Θα πρέπει να φροντίσουμε ε, οι πολίτες ε, να έχουν κριτικό πνεύμα. Ακούσαμε τις απόψεις των αρμοδιών επιτροπών και τώρα θα ακούσουμε τις απόψεις των πολιτικών ομάδων για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο κύριος Μπούζα, μισή λεπτό. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. ο πίτροπος έχει δίκιο συζητήσαμε για την εφαρμογή του προγράμματος με ένα πολύ φιλόδοξο τρόπο και μάλιστα όσο το δυνατόν ταχύτερα. Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία η ταχύτητα, αν υπάρχουν χρήματα για την κοινωνική κοινοτο... κοινο... καινοτομία, ε, ας πούμε την ιατρική η οποία είναι σημαντική. Θέλουμε να φτάσουν οι πόροι αυτοί εκεί όπου χρειάζονται το ταχύτερο δυνατό, δηλαδή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην έρευνα. Στο πλαίσιο, σε αυτό το πλαίσιο προγράμματος πρέπει να το θεσπίσουμε αυτό. Έχουμε το θέμα των αποστολών. Είναι μια πολύ καινοτόμο και εξαιρετική προσέγγιση. Ευχαριστούμε την Επιτροπή γιατί θέλουμε να καταλάβουν οι πολίτες τι σημαίνει πόλη με μηδέν εκπομπές ή η αντιμετώπιση του καρκίνου. Άρα είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, το οποίο θεσπίζει το πρόγραμμα, να είναι επιτυχημένο στο μέλλον όπως ως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Γιατί μην ξεχνάμε όλα τα πράγματα που θα πρέπει να μην μας διαφεύγουν. Είναι επίση σημαντικό να διευρυνθεί το πρόγραμμα στο βαθμό που είναι δυνατόν με την ανάπτυξη ειδικών πόρων για τα κράτη-μέλη. Όπως ας πούμε η Πολωνία, η οποία δεν χρησιμοποιεί πολύ τον ορίζο, το πρόγραμμα ορίζων μέχρι τώρα. Πρέπει να το προωθήσουμε. Ευχαριστώ λοιπόν τον Επίτροπο, την Ρουμανική Προεδρία, συγχαρητήρια, όπως επίσης και τους συναδέλφους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ για την ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών. Καπεσμό Ρουίζα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Με τον ορίζοντα Ευρώπη έχουμε τη νέα φιλοδοξία για να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Ε, χωρίς αποκλεισμούς. Γι' αυτό θα πρέπει να μετρήσουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο, όχι μόνο τον οικονομικό. Η επιστήμη θα πρέπει να λύσει τις προκλήσεις και τις αδικίες και να μην τις εντείνει και τις ανισότητες. Η Ευρώπη χρειάζεται όλα τα ταλέντα και τις γυναίκες. Γι' αυτό έχουμε μια ειδική ε, γραμμή στον προϋπολογισμό. Θα πρέπει να μειωθεί και ε, το χάσμα ανάμεσα στις περιφέρειες τα κλάστερ, να ενισχυθεί η υγεία, ε, κατά πολέμης κλιματικής αλλαγής, ψηφιακά, δημιουργική οικονομία, γαλάζια οικονομία και πάει λέγοντας. Θέλω όμως να τονίσω και το ρόλο που θα πρέπει να δοθεί στις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις, το 99% θα πρέπει να μειωθεί ε, το χάσμα της καινοτομίας της μικρομεσαίας. Θέλω να συγχαρώ όλη την ομάδα και το Επιτελείο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έκανε πραγματικότητα αυτό το σπουδαίο έργο. Ευχαριστούμε για την ομάδα ECR ο κύριος Τόσενόφς και μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές ήταν τεράστιε οι προσπάθειές τους και άριστη η συνεργασία τους με τους κοιότητε συζητητές και του ευχαριστώ γι' αυτό. Το Horizon Europe για την περίοδο 2021-2027 θα είναι ένα ισχυρό εργαλείο που θα ενισχύσει την έρευνα και την καινοτομία και θα βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, όχι μόνο στην ακαδημαϊκή έρευνα. Χαίρομαι που καταφέραμε να βρούμε ένα, να έχουμε μια κατάληξη ισορροπημένη παρότι δεν είχαμε πολύ χρόνο. Χαίρομαι επίσης που οι προτάσεις μου για τις ε, περιοχές του άνθρακα, όπως τις ονομάζω, ενσωματώθηκαν στην ε, πρόταση. Ήταν σημαντικό αυτό για να επιτύχουμε τους ενεργειακούς μας στόχους που έχουμε θέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Horizon Europe ε, θα διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και ειδικευμένων γνώσεων με κοινωνικές επιχειρήσεις, με ακαδημαϊκά ιδρύματα και με όσους ε, ασχολούνται με την εξόρυξη άνθρακα. Πρέπει να βελτιώσουμε την ανταλλαγή γνώσεων σε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι ο μόνο τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την ακαδημαϊκή γνώση και να σταματήσουμε τη διαρροή εγκεφαλών. Η κυρία για 1,5 λεπτό από του φιλελευθέρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε το ε, ένατο πρόγραμμα ε, πλαίσιο για την έρευνα και το συζητήσαμε εκτενώς και αύριο είναι κρίσιμη η ψηφοφορία. Αν εγκρίνουμε σε πρώτη ανάγνωση τον ορίζοντα Ευρώπη, θα εξασφαλίσουμε τη συνέχεια για τους επιστήμονες και τις καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία που έχω για να σας πω πόσο μοναδική είναι αυτή η ψηφοφορία. Μαζί με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς στο Κοινοβούλιο ε, πετύχαμε τα κατόρθωτα και τα διανόητα στον ε, τριμερή διάλογο. 18 μήνες ήταν η διαπραγμάτευση για τον ορίζοντα 2020, ενώ τώρα χρειάστηκε μόλις ένα τετράμινο. Αυτό είναι χάρη στην επικοδομητική συνεργασία και την κατανόηση που έδειξαν και τα τρία θεσμικά όργανα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερο τον Επίτροπο Κάρλος Μοέδας και ολόκληρο το επιτελείο του ε, που στάθηκε στο πλευρό μας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Εκτός αυτού θέλω να ευχαριστήσω και τους διαπραγματευτές της Ρουμανικής Προεδρίας. Η Ρουμανική Προεδρία είναι ισχυρό παράδειγμα για το πώς μπορούν και οι μικρότερες χώρες να παίξουν σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη. In για τους Ευρωπαίους πολίτες, για το μέλλον μας, για την έρευνα και την καινοτομία και στην επόμενη θητεία θα εξακολουθώ να πιέζω και να ζητώ 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ όμως απευθύνω έκκληση σε όλους να εγκρίνουμε αυτή τη σημαντική συμφωνία. Ευχαριστούμε Ματίας, εκ μέρους της για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τους συζητητές ε, για τις προσπάθειές τους κατάφεραν να ενσωματώσουν τις προτάσεις ε, τροπολογιών όλων των βουλευτών. Ευχαριστώ και την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τη διαπραγμάτευση αυτού του θέματος. Μας επέτρεψαν να καταλήξουμε σε καλή συμφωνία. Έρευνα και ανάπτυξη λοιπόν χωρίς αποκλεισμούς ε, ευρείες ε, με καινοτομία ως αποτέλεσμα. Καινοτομία όμως δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς βασικές γνώσεις, χωρίς τις κοινωνικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Είναι ένα συμβιβασμό, συμβιβασμού, συμβιβασμού. Κάτι λοιπόν που δεν είναι τέλειο Όλοι μας ε, θέλαμε να βάλουμε κάτι ουσιώδες ώστε να καταλήξουμε σε ένα συλλογικό αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω στις κοινωνικές επιστήμες, στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ίση πρόσβαση στα κονδύλια για όλους. Έχουμε έναν στόχο, ωστόσο όσον αφορά την έρευνα και όσον αφορά την έρευνα για την κλιματική αλλαγή. Το πρόγραμμα αυτό είναι το καλύτερο που έχει επιδείξει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οποιο γνωρίζει τους ερευνητές μας ξέρει τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να πω ότι οι υπεύθυνοι για αυτή την επιτυχία βρίσκονται κρυμμένοι στην τελευταία γραμμή, αλλά τους ξέρουμε όλους. Για τους πράσινου. ανταλύνετε για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εδώ και 50 χρόνια έχουν περάσει από τότε που πάτησε στο φεγγάρι ο Νίλ Άμστρονγκ το 1969. Ήταν ένα τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα. Ε, ήταν όμως και το αποτέλεσμα μιας αποστολής θαραλέας ε, και πολιτικού θάρρους. Το αντίστοιχο στη δική μας γενιά είναι η έρευνα στο ίδιο επίπεδο. Αυτό κάνουμε εδώ. Και αυτό θα ψηφίσουμε αύριο το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία. Ε, Εκτενεί διαπραγματεύσει και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω του συναδέλφου και τον Επίτροπο. Ποια είναι τα διακυβεύματα. Πρέπει να εξοπλιστούμε με καλύτερα μέσα για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές προκλήσεις. Εφόσον τα κονδύλια επαρκούν, θα έχουμε δισεκατομμύρια σουηδικέ κορώνες ε, για την πράσινη κινητικότητα, για την ε, πράσινη βιομηχανία. Και έτσι θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Ευχαριστούμε. Εκ μέρου του EFDT, ε, Ανταμάτο παρακαλώ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Σκιώδης Είμαι ικανοποιημένη και από τι δύο εκθέσει. Καταφέραμε να βρούμε μια καλή ισορροπία μεταξύ δραστηριοτήτων έρευνα και κοινοτομία. Πιέσαμε και ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Υποστηρίξαμε τον εγκάρσιο χαρακτήρα και τη συμπερίληψη των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών σε όλε τι δραστηριότητε του προγράμματο. Επιπλέον, εγγυηθήκαμε επαρκή υποστήριξη όχι μόνο στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα και στι startup, αλλά και στι μικρομεσαίε επιχειρήσεις με ένα ειδικό εργαλείο για αυτές. Έχουμε απογοητευτεί επειδή δόθηκε ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα που ακόμα περιορίζεται από την υπεράσπιση ιδιωτικών συμφερόντων και είμαστε δυσαρεστημένοι επειδή δεν δόθηκε επαρκή σημασία στην έρευνα για την ανάπτυξη. Όσον αφορά τη δομή της απόφασης, οι τομείς παρέμβασης ε, στον πυλώνα παγκοσμίων προκλήσεων και βιομηχανικής ε, ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, θα μας επιτρέψουν να παρεύουμε στην υγεία, στη δομή, στην ασφάλεια συμπεριλαμβανομένων των φυσικών καταστροφών αλλά και στη βιομηχανία, στο κλίμα, στην ενέργεια και στην κινητικότητα, στα προϊόντα διατροφής, στους φυσικούς πόρους, ε, στη γεωργία και στο περιβάλλον, ούτω ώστε να βελτιώσουμε την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Οι εργασίες για το Horizon Europe θα πρέπει να ολοκληρωθούν στην επόμενη θητεία αλλά όσα έγιναν μέχρι στιγμής ε, συγκεντρώνουν τα βασικά στοιχεία για την υποστηρίξη και την απαραίτητη πλαισίωση ώστε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας μέσω της έρευνας και της καινοτομίας. Ε, ευχαριστούμε. Κέλλη, ξεκινάει η συζήτηση. Κέλλη για 1,5 λεπτό. Χαίρομαι που μετά από τις σκληρές διαπραγματεύσεις ότι μπόρεσαν οι, οι να καταλήξουν σε συμφωνία για το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπης. Ευχαριστώ τους ε, συγητές, συγχαρητήρια και σε εσά Επίτροπε. Πραγματικά όλοι σας συγχαίρουν για αυτή την καλή δουλειά. Το πρόγραμμα αυτό θα στηριχθεί στα επιτεύγματα κάποιων πρόσφατων προγραμμάτων όπως ορίζουν 2020 και το FP7 για τη δημιουργία θέσεων εργασίας κυρίως στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, παραγωγής τροφίμων και άλλα. Αυτό είναι μια, ένα πολύ φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα, το πιο φιλόδοξο που ενισχύει την ε, δυνατότητα στον χώρο της επιστήμης και της έρευνας. Ε, ε, υπάρχει προπολογισμό που δόθηκε στο θέμα των τροφίμων και τη και αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να υπάρξουν ε, υγιή τρόφιμα τώρα και στο μέλλον ενώ υπάρχουν ε, αλλαγές στην αγορά και οι, αγο... καταναλωτές ζητούν τεχνολογικές εξελίξεις. Η παραγωγή τροφίμων θα είναι πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική στο παγκόσμιο περιβάλλον και θα, προσφ... θα καλύπτει διάφορες ανάγκες. Επίσης ε, υπάρχει ε, στήριξη στην, κλιματική, στην ενέργεια για την κλιματική αλλαγή και την έρευνα κατά του καρκίνου. Αυτό είναι εξαιρετικό κείμενο που θα, με χαρά θα υπερψηφίσω αύριο ε, και περιμένουμε να γίνουν και άλλα στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Πατρίτσια Τόια, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η συμφωνία για το Horizon είναι καλή είδηση για τους Ευρωπαίους πολίτες σίγουρα. Στο μέλλον θα έχουμε ένα πιο πλούσιο, πιο αποτελεσματικό, πιο απλό πρόγραμμα έρευνα, ελπίζουμε, και πιο διαφανέ. Σίγουρα θα δίνει μεγαλύτερη προσοχή στι οικονομικέ και κοινωνικέ επιπτώσει, όπω υπογραμμίστηκε, και θα δίνει προσοχή στην καινοτομία. Για το άνοιγμα αυτού του κεφαλαίου καινοτομία πρέπει να επενέσουμε τον Επίτροπο Μοίντα. Να συγχαρώ τον Νίκ, τον Έλερ και του ε, Καπεζών ε, σκιώδη ε, για τη δεσμευσή του. Πιστεύω ότι θα έχουν μεγάλη επιτυχία τα προγράμματα αυτά. Πρέπει να πούμε ότι εδώ η Ένωση μας ενδυναμώνει να αντιμετωπίσουμε κλιματικά προβλήματα που μια χώρα μόνη της δεν θα μπορούσε καν να αγγίξει. Είμαι ικανοποιημένη λοιπόν από την υποστήριξη που δίνεται στο νέο πρόγραμμα για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής και της ιταλικής οικονομίας Και το εργαλείο για τις ΜΜΕ πρέπει να συνεχιστεί στο Horizon και στο μέλλον, διότι έχει δώσει καλά αποτελέσματα. Ε, κάτι να θυμίσω για τις προτεραιότητες. Την υγεία, βασικό στοιχείο για τη ζωή των πολιτών και το κλίμα. Σήμα ακούσαμε την Κρέτα και πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσουμε ένα καλό μέλλον για τους νέους είναι να δεσμεύσουμε το μέγιστο ποσό πόρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των δυσκολιών που μας θέτει. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κρασνοδέψκη για ένα λεπτό. Θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές που κατάφεραν να, επιτύχουν συμφωνία στο θέμα στο, επί του ορίζοντα Ευρώπη. Ε, είναι δικαιολογημένε να τα συγχαρητήρια, γιατί αρχικά οι θέσεις του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου απήχαν πολύ μεταξύ τους. Μου άρεσε όμως καλύτερα η αρχική θέση του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Νίκα, ο εισηγητής, δικαιολογημένα υπογράμμισε την ανάγκη ε, να ε, προχωρήσει το θέμα της έρευνας. Όμως νομίζω ότι οι καταληκτικές προτάσεις, η, διεύρυνση συνεργασίας και το πακέτο δεν το καλύπτουν αυτό. Ανησυχώ ότι αυτό δεν θα μεταφραστεί σε απευθείας. Ε, εδώ ο συνάδελφος μιλάει στο τηλέφωνο μπροστά μου. Σας παρακαλώ, ζητήστε από, το, από τον ε, συνάδελφο να μην μιλάει στο τηλέφωνο. Αυτό φοβάμαι λοιπόν ότι δεν θα μετατραπεί σε πραγματική συνεργασία μεταξύ εταίρων ε, Κοιτώντα λοιπόν προς το μέλλον Θέλουμε ένα σχέδιο ώστε οι χώρες να μπορούν να βγουν από αυτό το συγκεκριμένο πακέτο. Μια λύση γι' αυτό είναι να συμπεριληφθεί συγκεκριμένος στόχος ποσοστών στον προϋπολογισμό για τις χώρες που συμμετέχουν στο διευρυμένο αυτό πρόγραμμα. Αυτό συμβαίνει σε διάφορα προγράμματα τώρα και κατά την υλοποίηση ελπίζουμε ότι η Κομισιόν θα φτιάξει ε, εφαρμοστικούς κανονισμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σταμπορένο, Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα αποτελέσματα. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για το 35% των δραστηριοτήτων που αφιερώνται στο κλίμα, την προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην πολιτιστική κληρονομιά, στις κοινωνικέ και Ανθρωπιστικέ προτεραιότητε. Ήθελα να απευθύνω μια έκκληση, καθώ κλείνουμε τη θητεία, ε, πολιτική έκκληση για λίγα λεπτά. Ο ανθρώπινο πολιτισμός πάντα χαρακτηριζόταν από τεχνολογική καινοτομία, από τα πρώτα βέλη, από το άρωτρο. Ο άνθρωπος πάντα χρησιμοποιούσε την τεχνολογία για να βελτιώσει τη ζωή του. Ωστόσο, από την άλλη, καινοτομία δεν έφερε πάντα βελτιώσεις οι Σουμέροι ανακάλυψαν ότι το σύστημα άρδευσή του αύξανε την αλατότητα των εδαφών και τα έκανε λιγότερο έφορα. Η βιομηχανική επανάσταση με τον άνθρακα έφερε τεράστια εξέλιξη αλλά έκανε τις πόλεις ανθυγιεινές και η μαζική κινητικότητα ε, δεν είχε προβλέψει την συμφόρηση στις πόλεις. Σήμερα έχουμε την ψηφιακή εξέλιξη που καθιστά δυνατό κάτι που παλιότερα θεωρεί το ε, ε, φαντασία. Ωστόσο, βλέπουμε οι αλγόριθμοι με τι συναλλαγέ υψηλή ταχύτητα, ε, ο έλεγχο τη ζωή, τη προσωπική ζωή των ατόμων, όπω γίνεται στην Κίνα, είναι από τα κακά αποτελέσματα. Και ε, ποιο μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη είναι καλύτερο να προλαμβάνουμε παρά να διορθώνουμε γιατί αργότερα είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως την πυρηνική απειλή, την κλιματική αλλαγή. Χρειαζόμαστε περισσότερη σοφία. Ε, ο καθένας να υπερασπίζει το δικό του κλάδο, ώστε ο καθένας να διατηρεί την αξιοπρέπειά του, την ψυχολογική και σωματική του υγεία, την ε, καθαρότητα των οικοσυστημάτων. Όλα αυτά θα πρέπει να βρισκόνται στο επίκεντρο οποιασδήποτε νομοθετικής ε, και βιομηχανικής εξέλιξης. Η επιστήμη πρέπει να υλοποιείται, αυτό είναι σημαντικό πάντα, χωρίς να ξεχνάμε τι μας έχει δώσει η φύση, μια φυσική ε, ευφυΐα σε ένα αναλογικό σώμα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε νου γη ενσώματη υγιή στο μέλλον και να ζούμε σε έναν ασφαλή πλανήτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κουντρίτσκα, παρακαλώ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς και είναι ακόμα πιο σημαντικό σε αυτούς τους καιρούς να ακούγεται δυνατά η φωνή της έρευνας, να βρισκόμαστε στην πλευρά μιας ισχυρής και συνεκτικής Ευρώπης που στηρίζεται στη γνώση και όχι στο λαϊκισμό. Πιστεύω ότι ο ορίζον Ευρώπη θα μας παράσχει αυτή τη δύναμη. Τα χάσματα στο χάρτη της Ευρώπης πριν από τον ε, ορίζοντα 2020 ήταν υπαρκτά. Το χάσμα αυτό τώρα γεφυρώνεται. Δεν έχω είναι υποχρεωτικό να υπάρχει Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Αυτό το νέο ερευνητικό πρόγραμμα θα δώσει προϋπολογισμό για την διεύρυνση της συμμετοχής στην έρευνα στις χώρες που δεν έχουν την τεχνογνωσία ή ισχυρή ερευνητική παράδοση. Θα μας επιτρέψει να εκπαιδεύσουμε εξαιρετικούς ερευνητές άσχετα από το ποια χώρα προέρχονται. Αυτό από μόνο το αποτελεί ανταμοιβή και είναι σαφής ένδειξη ότι η ευρωπαϊκή έρευνα είναι ισχυρή όταν όλη η Ευρώπη συγκεντρώνει συγκεντρώνει τις δυνάμεις της. Όταν έχουμε το 7 πρόγραμμα ε, πλαίσιο, επικεντρωνόμαστε στο ταλέντα της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Με το ε, νορίζοντα 2020 είχαμε την ιδέα να διευρύνουμε την τεχνογνωσία, αλλά δεν τα καταφέραμε πολύ γιατί είχαμε μόνο ε, 1% του προϋπολογισμού. Τώρα ορίζοντα Ευρώπη μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερο για στην γνώση στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην χρειάζεται να, βρουν τη δουλειά, ε, ε, να φύγουν τη χώρα του να βρουν δουλειά. Ευχαριστώ λοιπόν του συζητητέ, ευχαριστώ όλου, καθώ και την Ρουμανική Προεδρία. Τίποτα όμω δεν γίνονται εκ του μηδενών. Στρέφομαι λοιπόν στου πολιτικού. Στη νέα περίοδο μην περιμένετε τι μεταρρυθμίσει, εξυγχρονίστε τα πανεπιστήμια, χρησιμοποιήστε καλά τη διετία για να κάνετε καλή δουλειά. Μην ε, φύγετε από αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει. Κυρία Νίμπλερ, για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Και να σεβόμαστε τους χρόνους μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, αξιότιμε Προεδρεύων. Ποιο είναι το κλειδί για ένα επιτυχημένο μέλλον. Οι επενδύσεις, η καινοτομία και η έρευνα. Και συγχαρητήρια γιατί ήταν μαμούθ όλο αυτό το γιγάντιο έργο. Αγαπητοί φίλοι, με εσά κύριε Νίκα, με εσά κύριε Έλερ, με εσά κύριε μοετα και το Συμβούλιο, σε τόσο λίγο χρόνο καταφέραμε να δρομολογήσουμε 120 δισεκατομμύρια για την προαγωγή και τι επενδύσει στην έρευνα και ε, την καινοτομία. Σωστά είπε ο Επίτροπος Μοέτα ότι ε, βγάλαμε φωτογραφία τη μαύρη τρύπα στο Μόναχο ήμουν το Σαββατοκύριακο ε, στη μεγαλύτερη έκθεση ε, μηχανημάτων ε, κατασκευών και έχουν γίνει τεράστια άλματα για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία, τη νέα τεχνολογία και να βάλουμε τα θεμέλια για να ενισχύσουμε και τη βιομηχανία και ε, την έρευνα και στην υγεία και τις μεγάλες ασθένειες της εποχής που είναι ο καρκίνος και ε, ε, νόσος Alzheimer. Πραγματικά χαίρομαι πολύ και αν εγκρίνουμε το πρόγραμμα αυτό θα έχουμε στείλει και το σωστό μήνυμα για το μέλλον. Είναι εξαιρετικά τα μυαλά που έχουμε σε όλα τα κράτη-μέλη και το τονίζω σε όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να ενισχυθούν οι επενδύσει στην έρευνα και την καινοτομία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ κύριος Γκαμπούς για μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αυτή είναι η τελευταία μου παρέμβαση εδώ στο Κοινοβούλιο ως βουλευτής ε, μιλώ και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να τοποθετηθώ ακριβώς για αυτό το θέμα, Ορίζον Ευρώπη, γιατί συνοψίζει και τη δράση μου σε όλη αυτή τη θητεία. Βάζει τρεις μεγάλες προτεραιότητες κλειδιά από το νέο πρόγραμμα Ορίζον για να εξασφαλίσουμε καλύτερο μέλλον στις επόμενες γενιές. Κατά πολέμης κλιματικής αλλαγής, ψηφιακή οικονομία και υγεία. Σήμερα ακούσαμε πραγματικά τα συγκινητικά λόγια της Γκρέτα Τούμπερκ στην συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και επανειλημμένα την παραθέσαμε εδώ. Θα πρέπει να δράσουμε επιγόντως είναι απολύτω απαραίτητο κατά τη κλιματική αλλαγή. Δεν είναι επιλογή. Θα πρέπει η Ευρώπη να δίνει το καλό παράδειγμα και στο μέλλον, περνώντα από τα ε, λόγια στα έργα. Από εδώ λοιπόν προτείναμε το 35% των κονδυλίων του προγράμματος να ε, αφιερωθούν σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και μάλιστα περισσότερα προτείναμε εμεί από την Κομισιόν στην αρχή. Το δεύτερο, ψηφιακή οικονομία για να εξακολουθήσει να είναι η Ευρώπη πόλος έλξης γνώσης και ε, επιστήμης παγκοσμίω. Είναι το πρώτο πρόγραμμα, το μεγαλύτερο, για να εγγυηθούμε την ανεξαρτησία μας, δεν μπορούμε ε, ούτε επιτρέπεται να αφαιθούμε στα χέρια άλλων κάπως είναι οι γίγαντες της Ασίας ή οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και τέλος χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα για την υγεία, για την καταπολέμηση του καρκίνου και του παιδικού καρκίνου, χωρίς να ξεχάσουμε την έρευνα σε σπάνια νοσήματα και νοσήματα ψυχικής υγείας που επηρεάζουν χιλιάδες και εκατομμύρια Ευρωπαίων. Ευχαριστώ πολύ, ε, Επίτροπε. Και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και στα καταλανικά. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό κύριο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Δύο πράγματα θα ήθελα να τονίσω μόνο. Ακούσαμε πολλά για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του κλίματος και δεν μπορώ παρά να τα υπογραμμίσω. Σε αυτό όμως το πρόγραμμα Έχουμε πολύ ειδική στόχευση ε, για ε, την βιομηχανική παραγωγή ε, χωρίς διοξίδιο του άνθρακα. Είναι σημαντικό όταν το συζητούμε για την Ευρώπη και το κλίμα. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αποτελέσουμε το παράδειγμα παγκοσμίω. Οι Κινέζοι και οι Ινδοί δεν θα μας ακολουθήσουν αν έχουμε καταργήσει τα καυσαέρια και τις εκπομπές, αλλά να έχουμε καταργήσει και τη βιομηχανία. Γι' αυτό ε, εδώ και καιρό μελετούμε με τον Κρίστιαν Έλλαρ πώς θα μπορούμε για πρώτη φορά στην Ευρώπη να φτιάξουμε μια χαλιβουργία χωρίς διοξίδιο του άνθρακα. Το δεύτερο, ο καρκίνος, πολύ προσωπικό θέμα για όλους και για τον Μάνφρετ Φέμπερ, τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου μας, που μίλησε ήδη από το ε, Ελσίνκη για αυτό το θέμα όταν ορίστηκε υποψήφιος, γιατί έχασε τον αδελφό του από καρκίνο. Και έχουμε συζητήσει οι τρεις μας πολύ πώς μπορούμε να βοηθήσουμε άλλε οικογένειες για να μην έχουν να ζήσουν ε, ε, αυτή την πικρή εμπειρία. Ε, και έχουμε ασχοληθεί και με το θέμα του καρκίνου στα παιδιά, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ευτυχώς, δόξα το Θεό τα παιδιά αρρωσταίνουν σπανιότερα. Αλλά όταν αρρωστήσουν από καρκίνο είναι πάρα πολύ ε, σκληρό αυτό και πολύ οδυνηρό. Και μόνο ευρωπαϊκή συνεργασία μπορεί να βοηθήσει εκεί. Σα ευχαριστώ όλου και ιδιαίτερα τον Κρίστιαν Έλλερ, τον εισηγητή μα από το ΕΛΚ και σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε, Μπόνι, για ένα μισή λεπτό. Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Επίτροπε, θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές πολύ εγκάρδια για το επίτευγμα αυτό. Ορίζον Ευρώπη θα επιτρέψει για πρώτη φορά στην έρευνα να παίξει πραγματικό, συγκεκριμένο ρόλο στην πρόθεση, στην καθιέρωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Γι' αυτό πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε πλήρως το πρόγραμμα αυτό, ώστε να φτιάξουμε μια ε, ερευνητική έρευνα που θα στηρίζεται στην Ευρώπη, να, στηρίζ, να δημιουργήσουμε μια ερευνητική βάση και να συνδυάσουμε τους ιδιωτικούς πόρους με τους ευρωπαϊκούς πρέπει το πρόγραμμα να στοχεύσει κράτη-μέλη με, τα πιο αδύναμα αποτελέσματα. Είναι μια πολιτική συνοχής που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της Ευρώπης δύο ταχυτήτων. Η γνώση είναι απαραίτητο στοιχείο για την εξέλιξη. Χρειαζόμαστε ε, να έχουμε δια, διεπιστημονική, διαμεθοριακή, διακρατική συνεργασία για να τα πετύχουμε αυτά. Οι προϋποθέσεις αυτές μπορούν να μοχλεύσουν έξι φορές τις δυνατότητες των κονδυλίων και να προχωρήσουν χώρες που αυτή τη στιγμή δεν είναι ηγέτες στην Ευρώπη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας, ασφάλειας της ενέργειας, ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και να τα στρέψουμε προς την ε, εξυπηρέτηση ανθρωπότητας. Πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες ανάμεσα σε αυτό το πρόγραμμα, την πολιτική συνοχή, στα κοινωνικά ταμεία, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την εξειδικευμένη έρευνα. Η Πολωνία θέλει να ανεβάσει τον πύχη για, ε, στη χώρα γιατί ε, στην περίπτωση αυτή ο Ορίζον Ευρώπη θα βοηθήσει πολύ. Ευχαριστούμε Ζόφκο για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε Επιτρόπε, ως και εισηγήτρια για το Horizon Europe θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το ίδιο ισχύει και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Το πρόγραμμα Horizon Europe πρέπει να δημιουργήσει ευκαιρίες χρηματοδότησης δημιουργίας ε, και διατήρησης ε, κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Μπορούμε να ενισχύσουμε τους τοπικούς εφευρέτες και τους επιχειρηματίες ώστε να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Πρέπει να του ενθαρρύνουμε να παραμένουν και να αναπτύσσουν τις εφευρέσεις τους εκεί όπου βρίσκονται ώστε οι τοπικές κοινωνίες να υποφελούνται από τα επιτεύγματά τους. Η καλύτερη εικόνα είναι μια ιστορία ενός ε, Κροάτη επιχειρηματία Ματερή Μάτσα σε πρόσφατη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ε, ο επιτυχημένος επιχειρηματίας κατάφερε να δημιουργήσει ηλεκτρονικά συστήματα που έγιναν ε, φημισμένα σε όλο τον κόσμο, αλλά ε, αποτέλεσαν ε, και κίνητρο ανάπτυξης για την κροατική οικονομία δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασία. Μέσω όλων αυτών μπορούμε να εντείνουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ενδυναμώνοντας την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Φαρία, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, Καραμαέντας, Μαέντας, ε, αγαπητέ Μαέντας, ε, καλό απόγευμα. Θα θέλαμε να φέρνει καινοτομία αποτελέσματα, αλλά δεν φέρνει πάντα. Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν επιτευχθεί, δεν καταλήγουμε σε όλα τα αποτελέσματα που θέλουμε. Οπότε δεν μπορούμε να δεχθούμε μείωση τη χρηματοδότηση ε, του ορίζοντα και να υπερισχύσει η αρχή της προφύλαξης. Ε, κύριε Επίτροπε, ειδικότερα σε τομεί όπου χρειάζεται παρέμβαση, όπω για την καταπολέμηση τη χρήση του καπνού, ή τη χρήση ορισμένων χημικών προϊόντων στο γεωργικό και βιομηχανικό τομέα. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να εργαζόμαστε βάσει της αρχής της καινοτομία. Ε, που δεν αιτιολογείται. Πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στο κοινό συμφέρον για την υγεία με καινοτόμα προϊόντα. Είναι σημαντικό να έχουμε νέε επιστημονικέ έρευνε, αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των κινδύνων, των κόστων και των ωφελών. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορούμε να βρούμε νέες λύσεις ασφαλείς χωρίς να ζημιώνουν την υγεία των ανθρώπων. Ο Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Κάλιο αργά παρά ποτέ λέει μια παροιμία. άργησε η ευρωπαϊκή ένωση να καταλάβει ότι η ανταγωνιστικότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να στηριχθεί στην καινοτομία πρέπει να στηριχθεί στις νέες τεχνολογίες και όχι βέβαια στη μείωση των μισθών μια συνταγή την οποία επέβαλε στην ελλάδα επέβαλε σε πολλές χώρες του ευρωπαϊκού νότου. τώρα λοιπόν μιλούμε και πραγματικά πρέπει να προχωρήσουμε στις επενδύσεις γιατί μόνο με επενδύσεις στην τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπιστεί ο διεθνής ανταγωνισμός και ταυτόχρονα η τεχνολογία να μπει στην υπηρεσία του ανθρώπου να έχουμε παρεμβάσεις στα θέματα της υγείας να έχουμε φυσικά αναδιάταξη και της ίδιας της χαλιβουργίας για να μπορέσουμε να βλέπουμε μπροστά. όμως η τεχνολογία δεν μπορεί να είναι άλοθη για να γίνονται μαζικές απολύσεις. ετοιμάζουν 7.000 απολύσεις στην ελλάδα οι περίφημοι deutsche telekom η θυγατρική της δηλαδή ο ελληνικός οτε εν προκειμένου ο γερμανικός οτε. δεν μπορεί να ισχύσει αυτό κύριε επίτροπε στο όνομα της δίθεν ανάπτυξης τεχνολογίας μαζικέ απολύσει τι οποίες καταγγέλουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι στην ελλάδα. παρακολουθήστε το θέμα αυτό. Ζωρίνιο, παρακαλώ ένα λεπτό. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε αυτό το πρόγραμμα που είναι νέο, ε, το Horizon Europe με την ψηφιακή Ευρώπη θα ψηφιστεί σε αυτήν εδώ τη σύνοδο και θα φέρει ελπίζουμε αποτελέσματα. Χρειάζεται σύγκληση, ανταγωνιστικότητα και συνοχή. Κάθε χώρα πρέπει να κάνει βελτιώσεις ε, ε, εγχώριες ώστε να ωφεληθεί ολόκληρη η ευρωπαϊκή οικονομία, να υπάρχει μια συμμετρία θα ενισχυθούμε και εσωτερικά και στο να είμαστε πιο δυνατοί εσωτερικά θα εισακουστούμε περισσότερο εξωτερικά. Θα πρέπει λοιπόν ε, οι δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υλοποιηθούν με τρόπο αποκεντρωμένο. Όλα τα προγράμματα πρέπει να χαρακτηρίζονται από έναν κώδικα διοντολογίας προστασίας των αξιών ε, ε, που είναι ευρωπαϊκές. Και τέλος, ε, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και μετά το σημαντικότερο να έχουμε στο επίκεντρο όλων αυτών, όλης αυτής της έρευνας, ε, τον άνθρωπο. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, στον Επίτροπο. Είναι πολύ σημαντικό να ψηφίσουμε αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε. Ντάλι, παρακαλώ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα αυτής εξ αρχής να συγχαρώ και τους δύο εισαγητέ, αλλά και τον Επίτροπο για την θέσπιση του νέου προγράμματος πλαισίου πριν τις ευρωεκλογέ. γιατί πράγματι αυτό θα επιτρέψει την ομαλή υλοποίηση των μέσων χρηματοδότηση των διαδικασιών και των προϊόντων που εμπλέκονται. Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο αυτό έθεσε το θέμα της έρευνας και της καινοτομίας και του χάσματος ε, στην Ευρώπη πολύ σοβαρά. Είναι καιρός να ανοίξει αυτό το κλειστό ε, δίκτυο ε, στα κράτη-μέλη που έχουν χαμηλότερες επιδόσεις. Πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει ένα σύγχρονο, ε, μια σύγχρονη ανταγωνιστική και πραγματικά ανεπτυγμένη ε, οικονομία. Πρέπει να, χρησιμοποιηθεί τα υφιστά, να, ε, χρησιμοποιηθούν τα υφιστάμενα ερευνητικά ταλέντα και να προσελκυστούν νέα. Η ε, έρευνα και η τεχνολογία είναι θέμα κοινή ευθύνη και κάτι που πρέπει να το αναλάβουμε. Πρέπει να χαίρομαι που αναλαμβάνει ουσιαστική δράση η Ευρώπη από αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ το θέμα που δεν συζητείται εδώ σε όλη αυτή τη συζήτηση είναι φυσικά η θέση πολλών θεσμικών οργάνων του ε, Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν συμμετάσχει ιδιαίτερα στο προηγούμενο πρόγραμμα. Δεν φταίνε οι εισηγητέ ή οι διαπραγματευτέ, αλλά το θέμα του Brexit δεν έχει ακόμα επιληθεί. Παρά τα αυτά καθίσατε σαφέ ότι και ακόμα και αυτή η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα προσπαθήσει να συνεργαστεί στενά όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα του Brexit με το πρόγραμμα αυτό. Η μόνη απειλή είναι η ακραία το ακραίο Brexit που επιδιώκουν αυτοί που αρνούνται την κλιματική αλλαγή και οι λαϊκιστές. Παρά τα αυτά χαίρομαι ότι η ε, επιστημονική αριστεία παραμένει κριτήριο για την χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ορίζον. Ενισχύεται η έρευνα μέσω της συνεργασίας με την αριστεία. Ε, η, Ευρωπα... η παγκοσμίου επίπεδου ε, ερευνητική κοινότητα του Βασιλείου κάνει το πρόγραμμα ορίζον πιο επιτυχημένο. Ευχαριστώ πολύ. Κώστα, όχι δεν είναι εδώ. Τόμας, έτσι παρακαλώ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η καθιέρωση του Horizon Europe και των επιπλέον επενδύσεων για τις επιστήμες και την έρευνα αξίζουν επένους. Πρέπει να επενδύσει περισσότερα η Ευρώπη στις επιστήμες και στην καινοτομία για να γίνει παγκοσμία ανταγωνιστική. Σε αυτό το τομέα η Ένωση μπορεί πραγματικά να δείξει προστιθέμενη αξία, αλλά τα επιπλέον κονδύλια και η επιπλέον χρηματοδότηση δεν θα φέρει αποτελέσματα εάν δεν εκτιμηθούν ανάλογα με την αξία τους τα επιστημονικά επιτεύγματα. Είναι γνωστό ότι τα περισσότερα έργα που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο Έρευνας πάνε στα παλιά κράτη-μέλη, ενώ ε, τα νέα και λιγότερο αναπτυγμένα μέλη παίρνουν ψίχουλα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Παρομοίως, όλες οι χώρες του Horizon Europe πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα ανεξάρτητα από το που προέρχονται. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ελκύσουμε τους επιστήμονες ε, ε, να γίνουν καινοτόμοι, να παραμένουν στις χώρες τους και να δημιουργούν εκεί ευημερία. Ευημερία που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ολόκληρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέτερ, λέει, τελευταίος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στο έγγραφο αυτό υπάρχει και ένα κεφάλαιο που επιγράφεται «Χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια». Εγώ θα προτιμούσα να έλεγε «Χρειαζόμαστε περισσότερη υγεία», γιατί είναι ανησυχητικέ οι τάσεις. Οι μισοί πολίτες μπορεί να προσβληθούν από καρκίνο στην Ευρώπη. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερη Ευρώπη με λιγότερη υγεία και ε, ε, με περισσότερο καρκίνο. Η υγεία δεν είναι ένας κλάδος, είναι το μέλλον μας το ίδιο. Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο η υγεία παρά το Brexit που κάποια λύση θα βρεθεί. Το 70% των Ευρωπαίων επιθυμούν η Ευρώπη να δρά περισσότερο στα θέματα της υγείας και της πρόληψης. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα εκεί. Ως πρώην ασθενής καρκινοπαθής και πρόεδρος της ομάδας ε, της διακομματικής για την καταπολέμηση του καρκίνου. Ε, χαιρετίζω αυτή την ε, πρωτοβουλία να γίνει προτεραιότητα, μία από τις πέντε, το θέμα του καρκίνου. Ευχαριστούμε. Ο Επίτροπος Μέδας, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ θερμά αύριο μετά την ψηφοφορία μπορούμε να αρχίσουμε την προετοιμασία, τη δουλειά επί του στρατηγικού σχεδιασμού να δημιουργηθούν οι στόχοι και οι πρωτοβουλίες εταιρικής σχέση που χρειάζονται ώστε το 2021 το νέο πρόγραμμα ορίζων να έχει, είναι σε πλήρη λειτουργία. Αυτό ακριβώς κάνουμε σήμερα. Προετοιμαζόμαστε. Χαίρομαι πολύ. Είμαι πολύ περήφανος που βλέπω και αυτή είναι η τελευταία σύνοδος της 8ης νομοθετικής περίοδου. Σήμερα λοιπόν θα θυμάμαι, τη σημερινή μέρα θα τη θυμάμαι με πολύ ε, ευχαρίστηση γιατί όλοι από την αριστερά προς τη δεξιά, ο καθένας με τις διαφορετικές του ιδέες συνέκλινε. Συνέκλινε σε μια συμφωνία για το ότι πραγματικά μπορούμε κάτι να κάνουμε που θα αλλάξει τη ζωή των επιστημόνων, των ερευνητών και την ζωή και το μέλλον των παιδιών μας. Αυτή την καταπληκτική ανάμνηση θα την διατηρήσω. Σας ευχαριστώ όλους. Σε όλους όσοι βρίσκονται πίσω από από το προσκήνιο για όλα όσα έκαναν. Σας ευχαριστώ από βάθος καρδίας. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Τώρα το λόγο έχει ο εισηγητής ε, κ. Νίκα. Παρακαλώ, Ντάν, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο σήμερα και που είπαν ότι καταφέραμε να ενσωματώσουμε όλες τις προτάσεις ε, των μονιμών επιτροπών. Αυτό δείχνει ότι εντό του Κοινοβουλίου δείξαμε τεράστια ενότητα όσον αφορά το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κριστιαν Έλερ, τον συνάδελφό μου. Ε, συνεργαστήκαμε άρεστα. Ε, ευχαριστώ για το ανοιχτό μυαλό που έδειξε, τον πρέσβη επίση που μα βοήθησε να βγούμε από μια δύσκολη κατάσταση Κύριε Επίτροπε, τα τελευταία μου λόγια τα απευθύνω σε εσά. Ξέρω ότι η τωρινή Επιτροπή λίγη τον επόμενο Απρίλιο. Το καλό είναι ότι έχετε ένα χρόνο ακόμα και κατά το έτος αυτό θα σας ζητήσω εγώ κάποια πράγματα. Βεβαιωθείτε ότι το Horizon Europe δεν θα επηρεαστεί από τη γραφειοκρατία. Ας περικόψουμε τη γραφειοκρατία ώστε η έρευνα να ασχολείται με την έρευνα και λιγότερο με τη γραφειοκρατία. Μειώστε όσο το δυνατόν περισσότερο το διάστημα ε, ε, ε, που επιβάλλεται στους ερευνητές για την πρόσβαση και κάντε ό,τι μπορείτε για να βελτιώσουμε το πρόγραμμα αυτό να το αξιοποιήσουμε με την εκστρατεία ενημέρωση, ε, την υποστήριξη, γιατί χώρε όπω η Ρουμανία και οι άλλε χρειάζονται αυτή την ενημερωτική εκστρατεία. Όλοι πρέπει να ξέρουν πώ θα, πρέπει να ξέρουν πώς θα ετηθούν και ποιε είναι οι διαδικασίε. Τα ωφέλη θα είναι ε, θετικά για όλου μα. Ε, εγώ ελπίζω ότι θα συμμετέχω στο επόμενο κοινοβούλιο και από το φθινόπωρο και μετά θα φροντίσω να κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα. Διότι οι δικέ σα προσπάθειε, οι δικέ μου, των συναδέλφων μα, θα πρέπει να έχουν και πρακτικά αποτελέσματα άμεσα, αμέσω μετά από την αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστούμε για όλη σα την υποστήριξη. Ευχαριστούμε, κύριε Νίκα. Πάμε στον άλλο εισηγητή, κύριο Έιλερ, για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, επευκαιρία της απόψενής συζήτηση και της αυριανής ψήφισης του προγράμματος έρευνας, θα ήθελα να θυμίσω ότι η Ευρώπη έχει το θλιβερό ρεκόρ όπου ε, γεννήθηκε η ελευθερία της επιστήμης. Και μόνο εδώ πια διασφαλίζεται. Είναι μια νησίδα Στι Ηνωμένε Πολιτείε βγάζει φίρμα η κυβέρνηση να μην ερευνάμε για την κλιματική αλλαγή. Στην Κίνα, από την άλλη, ε, δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη ελευθερία έρευνα. Τότε θα πρέπει να τα θυμηθούμε και αυτά ε, με το ερευνητικό πρόγραμμα ότι ο αγώνας για την ελευθερία των επιστημών είναι από τους σημαντικότερους αγώνες που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η μάχη και σε παγκόσμιο επίπεδο και το ευρωπαϊκό παράδειγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για πάρα πολλού επιστήμονες παγκοσμίω. Και τέτοιες μέρε μέρες που ζούμε, μέρες Brexit, θα πρέπει να θυμούμε και ό,τι και να γίνει και με μεγάλη ενισχύα παρακολουθώ εκεί τις εξελίξεις, προφανέστατα το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ανήκει, γιατί ανήκει στην ερευνητική κοινότητα. Αν σκεφτούμε το Ηνωμένο Βασίλειο του περασμένου και προπερασμένου αιώνα ή του τωρινού. Από το 19ο αιώνα έχουμε αλληλεγγύη και συνεργασία με την Οξφόρδη, με το Κέμπριτζ και θα πρέπει να παραμείνει όσο γίνεται πιο κοντά μας στο Ηνωμένο Βασίλειο και ερευνητικά. Και τέλος, μετά τη συζήτηση αυτή, και όταν τελειώνει η θητεία, ο κάθε βουλευτής τίνει να ευλογάει τα γένια του. Και πολύ συχνά ακούμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι γραφειοκρατικό όργανο και αφηρημένο. Και θέλω να πω ότι ο Κάρλος Μοέδας πραγματικά τιμά με την παρουσία του το, ε, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έδειχνε μεγαλύτερη φιλοδοξία ο ίδιος πολλές φορές και ζήλο από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Και πραγματικά με χαρά εμείς κάπως συμπληρώσαμε αυτό το πρόγραμμα, αλλά είναι πραγματικά κοινή προσπάθεια και κοινό το επίτευγμα και με αποφυσικότητα τώρα ταινίζουμε το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Η κοινή συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά την έκθεση του κυρίου Ντάντι με θέμα εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων. Το λόγο έχει ο εισηγητής για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Επίτροπε Μπιανκόφσκα. Μετά από πολλά χρόνια και μετά από την αδικαιολόγητη διακοπή του νομοθετικού πακέτου για την ασφάλεια των προϊόντων του 2013, ήδη εγκρίνουμε νέου κανόνε για ένα σύστημα πιο αποτελεσματικό όσον αφορά του ελέγχου στην Ένωση. Ε, Ευχαριστώ. Χάρη στη συμφωνία, το Ευρωπαϊκό Σύστημα θα εξυγχρονιστεί, θα γίνει πιο αποτελεσματικό, πιο συντονισμένο. Θα διασφαλίζει ότι οι τελικοί καταναλωτέ ε, τελικά θα έχουν μπροστά του προϊόντα ασφαλή και συμμορφούμενα και ότι θα υπάρχει θεμητό ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά. Καθημερινά συναντάμε ε, παράνομα, παραποιημένα, επικίνδυνα προϊόντα. Όλο και περισσότερα. Κυρίω σε τομεί που επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα. Το 32% των παιχνιδιών, το 58% των ηλεκτρονικών συσκευών, το 47% των οικοδομικών προϊόντων δεν πληρούν τις βασικές προποθέσει ασφαλεία ή ενημέρωση προ του καταναλωτέ, όπω προβλέπει η νομοθεσία. Τα στα δεδομένα αυτά προστίθεται ο αυξανόμενος αριθμός παραποιημένων προϊόντων, πλαστών προϊόντων που πλήττουν ε, τις βιομηχανικές χώρες και αποτελούν αθέμητο ανταγωνισμό προς πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτά τα νούμερα και αυτές οι σκέψεις ε, μας οδηγούν στο να σκεφτούμε ότι είναι αποτελεσματικό το σύστημα ε, εποπτείας της αγοράς χωρίς επαρκή πόρους, χωρίς επαρκή συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ελάχιστη δυνατότητα αντίδραση ε, στι ε, παγκόσμιε ε, αλλαγέ. 500 είναι οι εθνικέ αρχές σε αυτό το σύστημα, αλλά δεν υπάρχει ούτε καν πλήρη χαρτογράφηση αυτών. Λείπει και αποτελεσματική επίσης επικοινωνία μεταξύ τους. Στην πρόταση της Κομισιόν, εμείς ως Κοινοβούλιο μελετήσαμε πολλά μέτωπα προσπαθώντα να ενσωματώσουμε κάποιε από τι προτεραιότητέ μα. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του κανονισμού είναι οι διατάξει που αφορούν του ε, φορεί αναφορά, όπω ονομάζονται, για τα περισσότερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη, τα πιο επικίνδυνα θα υπάρχει υποχρέωση να